Um, Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Νομικών Θεμάτων με την έγκριση της ημέρησης διάταξης. Έχουν γίνει εξή ε, αλλαγές στην αρχική ημερησία διάταξη. Στο σημείο 29 και 30 τα σημεία 29 και 30 μάλλον για την νομική βάση θα αναβληθούν. Το σημείο 32. Εξέταση μιας έκθεσης για τη διαδικασία μικροδιαφορών και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Πληρωμής θα αντιμετωπιστούν μετά το σημείο 41 που είναι η ψηφοφορία σε σχέση με την αναφορά 1784 κάθετος 2013. Έχετε κάποιες ε, αντιρρήσεις για την αλλαγή αυτή της ημερησίας διάταξης. Εάν όχι, η ημερησία διάταξη θεωρείται να ότι έχει εγκριθεί. Ανακοινώσεις Προέδρου, τίποτα δεν έχω να σας ανακοινώσω. Σημείο υπαριθμών 3. Η έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων της 3ης Σεπτεμβρίου, της 6ης Οκτωβρίου, της 13ης Οκτωβρίου και της 20ης Οκτωβρίου του ενεστώτος έτους, εάν δεν εγερθούν αντιρρήσεις προς τα πρακτικά, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Ως εκ τούτου, Μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο σημείο υπαριθμών 4 που είναι η ακρόαση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο. Στην προηγούμενη θητεία η Επιτροπή μας δημιούργησε μια ομάδα εργασία σε σχέση με το Διοικητικό Δίκαιο της οποίας, του οποίου μάλλον το, ε, της οποίας το έργο έληξε με μια έκθεση της οποίας ο εισηγητής ήταν ο Λίτζι Μπελίνγκουερ. Ένας ε, ιδιαίτερα εξέχων πρώην βουλευτής μέλος αυτής της Επιτροπής που χαίρομαι πάρα πολύ να τον καλωσορίσω και σήμερα πάλι. Η έκθεση αυτή συνοδεύτηκε από μια αξιολόγηση προστιθέμενης αξίας, ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, η οποία διεκρύβωσε ότι ένας ενιαίος, ένα ενιαίο διοικητικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνέβαλε τα μάλα σε μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή διοίκηση και θα έφερνε εξοικονομήσεις και συμβατά πρότυπα για το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το οποίο θα σήμαινε εξοικονόμηση χρόνου και μείωση άχθους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και φυσικά θα μείωνε και τις ε, ένδικες διαδικασίες, θα οδηγούσε σε καλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και θα οδηγούσε σε ορθολογικοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην τρέχουσα θητεία θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτήν την πρωτοβουλία ώστε να αφήσουμε και την Κομισιόν να κάνει τα απαραίτητα. Για αυτό το λόγο εμεί θα θα διορίσουμε ένα εισηγητή ο οποίος θα αναλάβει την σκητάλη από τον Λουίτζι Μπέρλιγκουερ. Εμείς έχουμε δύο ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι παρόντες εδώ σήμερα από την ομάδα Renewal, τους καθηγητές Χόφμαν και Σίδερ από τα Πανεπιστήμια του Λουξεμβούργου και της Παδίας. Χαίρομαι επίσης που μπορώ να καλωσορίσω την Dagmar Roth-Berendt, πρώην μέλος της Επιτροπής μας, η οποία ξέρει όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει κανείς για τη δημόσια διοίκηση και ιδίως την δημόσια διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία θα αναφερθεί στην πρωτοβουλία του Λουιζι Μπέλιγκερ και Μπελιγκουέρ και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μη καθυστερών περαιτέρω, θα δώσω λοιπόν το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, τον καθηγητή Χέρβικ Χόφμαν του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου. Ο καθηγητής Τσίρο θα, θα μιλήσει πρώτος. Εντάξει, έχετε το λόγο τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι εδώ μαζί με τον συνάδελφό μου Χόφμαν για να σας παρουσιάσουμε τις εργασίες μας σε μια ερευνητική ομάδα Renewal που λεγόταν και που είναι ένα πανεπιστημιακό δίκτυο που εδώ και πέντε χρόνια μελετάει συγκεκριμένα προβλήματα διοικητικού δικαίου, ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου και ιδιαίτερα η ομάδα αυτή συνέγραψε με ολόκληρη επιτροπή 15 μελή και από πάνω από άλλα 100 μέλη που, των οποίων τα ονόματα μπορείτε να τα βρείτε στο, στην μας συνέγραψαν κανόνες που εστάλησαν και σε εσά που υποβάλαμε από την 1η Σεπτεμβρίου. Οι κανόνες αυτοί εμφαίνονται σε μια μελέτη που εδώ και πέντε χρόνια είχε συνταχθεί και αναφέρονται σε ορισμένα σημαντικά σημεία όπως διασκέψεις που έχουν οργανωθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 12 και το 14 και μετά από τις ε, διασκέψεις αυτές συναντηθήκαμε και άλλες φορές με εμπειρογνώμονες από διάφορους κύκλους, υποδημοσίους υπαλλήλους, δικαστάς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή οργανώσεων πολιτών και υπάρχουν στα αγγλικά από την 1η Σεπτεμβρίου θα μεταφραστούν και στα ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και πολωνικά. Τώρα γίνονται οι μεταφράσεις. Η παρουσίασή μου θα επικεντρωθεί σε δύο ερωτήματα. Γιατί να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός διοικητικός κώδικας, γιατί στις λατινικές γλώσσες δεν μιλάμε για νόμο αλλά για κώδικα, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Και στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά όλα βέβαια που θα σας παρουσιάσω τα λέει πολύ πιο λεπτομερώς στο πρώτο βιβλίο των κανόνων στο οποίο θα αναφερθεί ο συντάδελφός μου Χόφμαν. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει την εισαγωγή αυτούς τους νέους πρότυπους κανόνες. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, γιατί να υπάρχει ένας τέτοιος κώδικας ή νόμος για το Ευρωπαϊκό Διοικητή, Ευρωπαϊκές Διοικητικές Διαδικασίες. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για τη μεταφορά των θεσμικών αξιών μας στην πραγματική ζωή των οργανισμών της Ένωσης και των υπηρεσιών της θεσμικές αξίες που είναι η προστασία του κράτους δικαίου, η νομιμότητα, η νομική βεβαιότητα, αναλογικότητα των ε, μέτρων κλπ. Ε, βέβαια θέλουμε μια ένωση δημοκρατική και διαφανή και άρανα και προστασία του δικαιώματος συμμετοχής και πρόσβασης στην πληροφόρηση και φυσικά και τις αρχές που έχουν καταγραφεί στο άρθρο 41 της Χάρτας των Θεμελιωδών και που αφορούν το δικαίωμα σε καλή και χρηστή διοίκηση. Ωραία, γιατί αυτός ο κώδικας διοικητικών διαδικασιών, ο λόγος, πέρα από τη μεταφορά των θεσμικών αξιών ή συνταγματικών αξιών, είναι ότι έγινε μια μελέτη υπό τον Λουίτζι Μπερλιγκουέρ και που από τη μεριά μας κάναμε και εμείς ως πανεκαδημαϊκοί και που έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός των υπαρχόντων κανόνων ως προς τις διοικητικές διαδικασίες που είναι οι κανόνες αυτοί κατακαιρματισμένοι σε διάφορες ειδικεύσει πολιτικές και υπάρχουν και διαδικαστικά στοιχεία που δεν επαναλαμβάνονται σε όλους τους τομείς άρα υπάρχουν μεγάλα ελλείψεις στους κανόνες της διοικητικής διαδικασίας στην Ένωση και όταν υπάρχουν ελλείψεις το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αναφερθούμε στις γενικές αρχές του δικαίου, αλλά μόνο το δικαστήριο μπορεί να μας πει τι είναι και τι δεν είναι γενική αρχή δικαίου. Και άρα και για τους ίδιους τους διοικητικούς και για το κοινό αυτό αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε ότι το καλό του υπάρχοντος συστήματος είναι ότι οι κανόνες που ισχύουν έχουν αναπτυχθεί, έχουν δημιουργηθεί και δυναμικά και πειραματικά. Γι' αυτό είναι διαφορετική ανατομία. Αυτό είναι καλό, αλλά έχει και τα μειονεκτήματά του. Και μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μερικά μαθήματα από την εμπειρία των χωρών μελών και από, άλλα τρίτε, από άλλες τρίτες ως προς την κωδικοποίηση της διοικητικής διαδικασία μαθήματα που προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όσο το δυνατόν καλύτερα στις εργασίες μας που βασίστηκαν μεταξύ άλλων και σε αναλύσεις σε πολύπλοκες νομικές αναλύσεις από τις διάφορες χώρες. Στην Ισπανία, ας πούμε, υπήρχαν παραδείγματα μιας πρώτης προσπάθειας κωδικοποίηση, μετά στην Αυστρία με πρώτη και δεύτερη φάση, στη Γερμανία επίσης το 1976 και ενδιαφερθήκαμε και, σε, και για άλλες περιπτώσεις όπως των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν έναν κώδικα διοικητικής διαδικασίας από το 1946 και στη Γαλλία υπήρχε μεγάλη αντίσταση στην ιδέα ενοποίησης ή κωδικοποίησης λέγω, έγανε αρκεί η κωδικοποιηση λεγω εγανε αρκει ώστε το δίκαιο να αναπτυχθεί από μόνο του με την ομολογία. Αλλά και σήμερα ακόμα, αλλά και σήμερα και ακόμα και στη Γαλλία γίνεται μια προσπάθεια κωδικοποίηση. Όλα αυτά τα πρότυπα είναι χρήσιμα, αλλά κανένα δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει. Το κύριο μάθημα που πήραμε από τις εργασίες μας είναι ότι αντίθετα από αυτό που λέγεται συχνά, αυτές οι κωδικοποιήσεις δεν κατέληξαν τελικά σε αύξηση των διαμαχών ή των συγκρούσεων. Γιατί η γνώση των αρχών αυτών απέφυγε αντίθετα τη δημιουργία διαφορών. διαφορών. Υπάρχει και ένα, μια, ένας τέταρτος λόγος υπέρ της δημιουργίας μια τέτοιας κωδικοποίησης που τον ανέφερε και ο πρόεδρος σας προηγουμένως η αξιολόγηση που έγινε από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έδειξε ότι υπάρχουν θέματα διατύπωση, προβλήματα διατύπωσης στις διάφορες γλώσσες, διατύπωσης που είναι δυσνόητη για το κοινό και για τον δημόσιο υπάλληλο που πρέπει να εφαρμόσει. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα νομικής βάσης. Για μας δεν είναι πρωτεύον αυτό το πρόβλημα, αλλά θελήσαμε να ασχοληθούμε και με αυτό για να είμαστε ρεαλιστέ. Διότι ξέρουμε ότι αν προτείνουμε στους νομοθέτες, στους νομοθέτη και στους θεσμούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το νέο κώδικα κάτι που δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κανονισμό της Ένωσης, τότε η δουλειά αυτή θα έχει γίνει τζάμπα και βέρεσε θα έχει μόνο ακαδημαϊκή αξία θεωρητική. Γι' αυτό θελήσαμε να δούμε και το θέμα των νομικών υποβάθρων και βάσεων και το βασικό που συζητήσαμε αφορούσε την εφαρμοσιμότητα ημί του άρθρου 198. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Ας μην υπησέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά τα προβλήματα αυτά του 298 με θεωρούμε ότι μπορούν να λυθούν εφόσον το περιεχόμενο των κανόνων είναι σαφές. Υπάρχει έπειτα ένα πολιτικό πρόβλημα, πολύ σημαντικότερο από το νομικό, του νομικού υποβάθρου και που αφορά το πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα όργανα και οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης ή μήπως να εφαρμόζεται και στις διοικήσεις των χωρών μελών όποτε αυτά εφαρμόζουν ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως τη Χάρτα των Θεμελιωδών. Η απάντησή μας είναι ότι από νομικής πλευράς και οι δύο απόψεις είναι θεμητές, αλλά από πολιτικής δεν θα ήταν ρεαλιστικό να θελήσουμε αμέσως να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε διοικητικούς κανόνες ομοιόμορφα από όλες τις υπηρεσίες και των χωρών μελών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι η συνεργα... θα ήταν η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών. Επιλέξαμε λοιπόν να πούμε το εξής. Γνωρίζουμε απολύτως ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε τη χρησιμότητα αυτού του κώδικα είναι να τους, του υποβάλουμε και να τους αναλύσετε κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να σας παρουσιάσω σήμερα κάποιες ιδέες που έχουμε αναπτύξει και που αν συμφωνήσετε μαζί μου απηχούν και το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ιανουαρίου 2013. ως συγκεκριμενοποίηση τελικά του συνταγματικού σας δικαίου. Αναφέρομαι σε τρεις ερωτήσεις. Είναι η σωστή χρονική στιγμή, όπως είπε και ο συνάδελφος μου πριν. Τελικά κωδικοποίηση ποιου πράγματος και ποια είναι τα μεγάλα υποφόσπαντα προβλήματα στο πλαίσιο αυτό. Το βασικό λοιπόν ερώτημα, γιατί άραγε θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο το πρόβλημα αυτό του διοικητικού δικονομικού δικαίου, είναι η σοβαρή ποικιλομορφία σε διάφορους τομείς που εμποδίζουν μια συνεκτική ανάπτυξη του διοικητικού δικονομικού δικαίου και την νομιμοποίησή του. Υπάρχει νομική βάση. Άρα πρέπει να εξετάσουμε τώρα πώς να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, την νομιμοποίηση και τη διαδικαστική νομιμοποίηση. Πώς λοιπόν να προχωρήσει άραγε κανείς. Μελετήσαμε διάφορες προσεγγίσεις από διάφορα νομικά συστήματα διάφορων χωρών μελών, αλλά και εκτός της Ένωσης και μας έδειξαν αυτές ότι η καλύτερη λύση είναι να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα, να δούμε δηλαδή τι είδους διαδικασίες υπάρχουν και να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία. Και αυτό μας οδήγησε να καταλήξουμε σε μια λίστα ενιών, εκτελεστική ε, διαδικασία, ε, απόφαση αναπερίπτωση, συμβάσεις και κάτι που το λέμε εμείς information management, δηλαδή αμοιβαία ε, παροχή βοήθειας, όπως για παράδειγμα στο Schengen. Τώρα για τη θέσπιση κανόνων, ποια είναι τα μεγαλύτερα θέματα εδώ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οι κανόνες μέσα στη συνθήκη για τις εκτελεστικές και καταξιότητες πράξεις, αυτές παραπέμπουν όμως στη συνθήκη, καθώς επίσης και στον κανονισμό επιτροπολογίας, και περιλαμβάνουν διαδικασίες για το τι θα γίνει μετά από την υποβολή της προτάσεως από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν εξετάζουμε την νομοθεσία στην οποία έχει συμβάλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μέσω των διαδικασιών μέχρι ότου έρθει η στιγμή όπου θα κατατεθεί πραγματικά η πρόταση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη συνοχής για το πώς να μεταφερθούν οι συνταγματικές αρχές στην πράξη και σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων πολιτικής. Εκεί υπάρχει μεγάλο δυναμικό απλούστευσης, όχι μόνο σε ειδική νομοθεσία, αλλά και για να υπάρξει διευκρίνηση, να υπάρξει διασάφηση. Εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία, αυτό που κάναμε με το, δίκαιο, με, συγγνώμη, με το δίκτυο μελέτης μας ήταν να το σπάσουμε, να σπάσουμε τα τμήματα σε διάφορα μέρη, να δούμε αυτό το rule making, ποιες βασικές αρχές έχει, και να αρχίσουμε, όταν αρχίζουμε δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα δημοσιοποίησης της πρόθεσης και του φάσματος εφαρμογής των όσων θέλουμε. Αν χρειαζόμαστε για παράδειγμα για και μελέτες αντικτύπου και για διοικητικά νομοθετήματα, τα οποία επίσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του πολίτη και μάλιστα ίσως και περισσότερο από την ουσιαστική νομοθεσία πώς επίσης θα γίνει διαβούλευση με τον επιστημονικό τομέα, πώς θα εξηγήσετε σε μια διασαφητική, σε μια εισηγητική έκθεση το σκοπό του νομοθετήματος. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την διαδικασία θέσπισης των κανόνων. Θεσπίζοντας λοιπόν τις σχετικές διαδικασίες μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι συνταγματικές αρχές θα είναι ορατές και θα τη ζει ο κόσμος καθημερινά. Ο δεύτερος ε, σημαντικός τομέας προβλημάτων των διοικητικών διαδικασιών είναι η απόφαση ανά υπόθεση, ανά περίπτωση, το οποίο γνωρίζουν όλα σχεδόν τα υπηρετικά ευρωπαϊκά συστήματα και είναι βέβαια και ο βασικός στόχος του άρθρου 41 που αναφέρθηκε και πριν. Στον τομέα αυτό πάλι ειδικά κατά τομέα υπάρχουν κανόνες πολύ συχνοί Πολύ συχνά λοιπόν διοικητικοί κανόνες ανατομέα. Αλλά το επίπεδο λεπτομέρειας είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει στάνταρτ προσέγγιση και γι' αυτό υπάρχει μεγάλο πλήθος περιττών περιπλοκών και υπάρχει σημαντική ανάγκη να διασαφηθούν οι κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και πάλι λαμβάνοντας την ίδια προσέγγιση, δηλαδή αναλύοντας την λήψη αποφάσεων στις διάφορες φάσεις της, βλέπουμε τους κανόνες στα εθνικά δίκαια, βλέπουμε και στις πολιτικές ανατομής της Ένωσης, που πρέπει, οφείλουν να περιέχουν θέματα του πότε γίνεται η αίτηση, πότε υποβάλλεται η αίτηση, πότε αρχίζει μια διαδικασία να τρέχει, προθεσμίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται, να δημοσιοποιούνται οι ε, εξουσίες διαρεύνησης που πρέπει επίσης να είναι γνωστές Χρειάζονται λοιπόν επίσης συγκεκριμένοι κανόνες που θα είναι κοινοί και για τη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και τις ευρωπαϊκές αρχές, διότι η λήψη αποφάσεων είναι ο τομέας του, του φαινομένου εκείνου της υποχρεωτικής αρμοδιότητας. Έχουμε δηλαδή χώρο όπου η αρμοδιότητα δεν ανήκει ούτε στη χώρα μέλος ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις δύο πλευρές. Και αυτό οδηγεί στην πραγματικότητα σε πολλά προβλήματα για τα μεμονωμένα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν εν τέλει ποιο είναι αρμόδιος και επίσης τα δικαστήρια δεν γνωρίζουν ποιο δίκαιο τυχαίνει να είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με την έννοια αυτή, τα θέματα αυτά λοιπόν απαιτούν την προσοχή μας όταν εξετάζουμε το rule making. Ο τρίτος μεγάλος χώρος που είναι οι συμβάσεις. Συνήθως αυτές συνδέονται με τις δημόσιες προμήθειες. Αν όμως ψάξει κανείς λίγο περισσότερο, διαπιστώνει ότι οι συμβάσεις είναι εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται μέσα σε όλο το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο, είτε για τη χρηματοδότηση της έρευνας, είτε για χρηματοδοτήσεις άλλων έργων, είτε για την επίλυση διαφορών, αλλά επίσης και για την υποστήριξη μονομερών αποφάσεων για παράδειγμα, μια απόφαση σχετικά μια συγχώνευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό ανακύπτουν και εδώ σημαντικά ερωτηματικά. Πρέπει το δημόσιο δίκαιο των συμβάσεων να μείνει στα γενικά ή πρέπει να εξειδικευτεί. Και οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να φροντίσουμε ώστε οι δημόσιες διοικήσεις να μην ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητές τους που τους επιβάλλει το δημόσιο δίκαιο μετακινούμενες στο συμβατικό δίκαιο, στο δίκαιο των συμβάσεων δηλαδή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την διερεύνηση, ακροάσεις, ε, διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς κλπ. Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν μέσα στο δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων. Και τέλος, στην ε, αμοιβαία συνδρομή, και αυτό είναι σημαντικό να νομοθετηθεί, διότι αν εξετάσετε τον κάθε ένα οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς δημιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία και έχουν συχνά την υποχρέωση να κάνουν κάποια ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και στα άτομα, όχι μόνο εκείνων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στα συστήματα, αλλά και τρίτων μερών που θίγονται από αυτή τη συνεργασία. Άρα λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με την προστασία δεδομένων και με την πρόσβαση της προφορίας στους τομείς αυτούς, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτή την έννοια της υποχρεωτικής αρμοδιότητας, διότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία οδηγούν στον συντονισμό των δράσεων των χωρών μελών με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και αυτή είναι η στιγμή όπου αρχίζει να γίνεται πια όχι τόσο σαφής η πραγματική ευθύνη, αρμοδιότητα. Θα τα εξετάσουμε αυτά, μάλλον μπορείτε να τα δείτε αυτά σε λεπτομέρεια στο υλικό που σας έχουμε διανύμει. Έχουμε τώρα τις μεγάλες ερωτήσεις. Την σχέση πρώτα, σχετικά με το εάν το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο εφαρμόζεται μοναχά σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, λειτουργού κλπ. ή και σε αυτό το χώρο μελών. Η απάντησή μα είναι ότι πολιτικά ξεκινά από το ένα, αλλά δεν λησμονεί και την υποχρεωτική αρμοδιότητα, compulsive procedures, υποχρεωτικέ διαδικασίε, όπου εκεί ε, μπαίνουν και στα χωράφια των χωρών μελών. Το άλλο θέμα είναι εάν οι διοικητικέ διαδικασίε κάποιου είδου αποφασίζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς συνδέονται με τις συγκεκριμένες αποφάσεις που λαμβάνονται στο, σε άλλα επίπεδα. Μπορεί κανείς να επιλέξει την ελάχιστη προσέγγιση ή να πει ότι ορθοί κανόνες θα πρέπει να έχουν και το ρόλο του υποδείγματος και ειδικέ ανατομέα πολιτικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι εξαιρέσει. Εμεί αποφασίσαμε λοιπόν ότι το καλύτερο είναι να μπαίνουν συνολικά οι κανόνε και θα να μπορούν να προβλέπονται εξαιρέσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. both... Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και του δύο καθηγητέ και για το γεγονό ότι παρέμειναν μέσα στο χρονικό τη ώρας. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο well. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Και θυμάμαι με πόσο ενθουσιασμό και με πόση χαρά έχω σταθεί μέλος της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες. Ξεκινώ λέγοντας ότι πρέπει να προωθήσουμε την ολοκλήρωση στο διοικητικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποκεντρωμένοι φορείς γίνονται σιγά σιγά ε, τμήματα μιας ενιαίας δομής σε πολλούς ε, χώρους και γίνεται εφικτό αλλά και ρεαλιστικό να δώσουμε την υποστήριξή μας σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο έργο η δικαστική αρρωγή και συνεργασία, αλλά γίνεται τώρα κάτι το απαραίτητο, γιατί το διοικητικό δίκαιο βασίζεται, όπως ελέγχθη, σε οικουμενικές αρχές. Είναι τμήμα της δημοκρατίας η διαδικαστική και οι κανόνες ουσιαστικού δικαίου θα πρέπει να προχωρούν παράλληλα. Δεν θα υπάρξει καμία ολοκλήρωση στην Ευρώπη χωρίς να παίξει το ρόλο του το δίκαιο το οποίο διέπει τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε όλο και σε πιο στενή και βαθιά ολοκλήρωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να βελτιώσουμε και το νομικό πλαίσιο. Η δικαστική συνεργασία είναι απαραίτητη και κέρια για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σύμφωνα με τις συνθήκες, οι διαδικασίες προδικαστικού χαρακτήρα εξασφαλίζουν την ενιαία ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Όχι μονάχα όμως με εθελοντική βάση, όταν γίνονται σε εθελοντική βάση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε και αρχές στο επίπεδο το ευρωπαϊκό για το διοικητικό δίκαιο που να ρυθμίζουν τις διοικητικές διαδικασίες. Η ανάπτυξη της νομολογίας είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε ένα επίπεδο επικουρικό και περιορισμένο. Είναι κέριος αυτός ο ρόλος. Στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησαμε με μία νομοθετικού χαρακτήρα έκθεση. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αποκομίσαμε κάποια επίπεδα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ώστε να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια απλή και σύντομη κωδικοποίηση των θεμελιωδών αρχών που θα πρέπει να ρυθμίζουν τη δράση των δημοσίων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείναμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να υποβάλει μια πρόταση κανονισμού σε σχέση με ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διοικητικών Διαδικασιών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου δεν εξαρτάται μόνο από τα νομοθετήματα, τους κανονισμούς, οδηγίες κτλ. αλλά και από την ομολογία που προκύπτει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τα άλλα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα της δράσης αυτών των δύο στοιχείων επί τη βάση των γενικών αρχών. Ορισμένες αρχές οι οποίες είναι ε, σχετικές με τις εθνικές διοικήσεις έχουν μεταφερθεί και έχουν αναπτυχθεί βαθμία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματα. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου σε σχέση με το διοικητικό τομέα δεν αφορά μονάχα την άμεση διοίκηση από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εθνικές διοικήσεις μέσα στο πλαίσιο αυτό και η νομολογία στην οποία έχω αναφερθεί προηγουμένως έχει κωδικοποιηθεί σε πράξεις δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η οδηγία περί παροχής υπηρεσιών. Πρέπει βάσει αυτών των νομοθετημάτων να δημιουργηθούν ε, ειδικέ αρχές όπως παραγωγικά μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην πράξη, οι εθνικές διοικητικές ε, δικαστικά δικαστήρια και δικαστικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν όλες αυτές τις αρχές και ιδίως τα δικονομικά δικαιώματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι η ισοδυναμία και η αποτελεσματικότητα στον τομέα του διοικητικού δικαίου. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε πια να πούμε παρά τις μακρές συζητήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί όταν έλεγαν όλοι ότι βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, ένα κράτος, μπορούμε πια να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο του να έχουμε ένα ενιαίο διοικητικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίκαιο. Και αυτό είναι και ο κύριος ρόλος για τον οποίο έχει σημασία αυτή η συζήτηση. Τα... <clears throat> Μπορεί να υπάρξει διοικητικό δίκαιο ακόμα και για οντότητες οι οποίες δεν είναι κρατικού χαρακτήρα. Η Κομισιόν αναφέρεται στην έννοια της διοίκησης που έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει τονίσει ήδη από την αρχή την ε, σημασία του να υπάρχει μια σχέση διοικητικού δικαίου όχι μονάχα με τα κράτη-μέλη αλλά και με τους πολίτες. Η περίπτωση Van and Laws όταν το δικαστήριο ανέφερε ότι τα υποκείμενα δικαίου δεν ήταν μονάχα τα κράτη-μέλη αλλά και οι πολίτες. Και υπάρχει το υπόδειγμα της συνδιοίκησης ή της ολοκληρωμένης διοικητικής διοίκησης. Επομένως, το ενωσιακό διοικητικό δίκαιο επηρεάζει και το διοικητικό δίκαιο των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος, τις εγγύησεις που παρέχουν. Επομένως, για, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η ενιαία δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχών του διοικητικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο έχει ορισμένες αρχές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αρχές οι οποίες έχουν ιονή συνταγματικό χαρακτήρα. Η σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ ο ευρωπαϊκός νόμος ε, ουσιαστικά συναρμόζεται με τον εθνικό νόμο. Οι νομολογίες οι οποίες προκύπτουν είναι και πάλι ένα ειδικό τμήμα της νομοθεσίας. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για διοικητική πολυμορφία, αλλά που υπόκειται σε εθνικές αρχές, σε, αρχές, ώστε να είναι αυτός ο πλουραλισμός συμβατός με τις γενικές ευρωπαϊκές αρχές. Όλα αυτά τα οποία έχουν λάβει χώρα μετά από την έγκριση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και μετά από την πρόσφατη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι έχουμε πια τμήματα δικαίου τα οποία έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και υποχρεώνουν τα κατημέλη σε συντονισμό των διοικητικών προσπαθειών τους. Ιδίως το άρθρο 298 όπως αναφέρθηκε, το οποίο αναγνωρίζει επίσημα την ύπαρξη διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χάρτα, το άρθρο 41, που αναφέρεται και στην έννοια της ε, υπηκότητος σε διοικητικό επίπεδο. Και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο με τη δημιουργία της ομάδος εργασίας, με τη λήψη υπόψη των ε, εκθέσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση από την Επιτροπή αυτή ομόφωνα και στη συνέχεια ενεκρίθη με ευρύτατη πλειοψηφία στην ολομέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης αποτελεί ένα δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και δίνει έτσι μια απάντηση στα αιτήματα για δημοκρατία, για διαφάνεια, για αναμονιμοποίηση. Γι' αυτό το λόγο <clears throat> χρειαζόμαστε ένα ε, διαδικαστικό διοικητικό δίκαιο. Και τώρα φυσικά η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει συνέχεια. Το τονίζω αυτό ειλικρινά. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε την Κομισιόν να κάνει κάτι το οποίο καταρχήν θα πρέπει να είναι δική της πρωτοβουλία. Να αντιμετωπίσει ακριβώς το έργο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και τα θέματα που συνάπτονται με τη διοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε μια απάντηση από την Κομισιόν η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια διαδικασία λεπτομερή για την αποτύπωση της νομικής πραγματικότητας στο διοικητικό τομέα και θα διακριβώσει αν υπάρχουν παραδείγματα ε, που να οφείλονται σε κενά ή σε ελλείψεις στο τωρινό νομικό πλαίσιο και επίσης θα εξετάσει το πώς θα μπορέσουν να αποφευθούν αντίστοιχα τέτοια προβλήματα στο μέλλον, ενδεχομένως με πιο συγκεκριμένη δράση κάποιου από τα θεσμικά μας όργανα. Αν εξετάσω τώρα το ύφος και τη γλώσσα, βλέπω να την διατρέχει την ε, δήλωση της Κομισιόν ο δισταγμός. Χρειάζονται αιώνες για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Θα πρέπει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και να αντιμετωπίσουμε και την πραγματική εφαρμογή του διοικητικού δικαίου. Αυτό όμως αποτελεί, αυτό απαιτεί μια πρωτοβουλία και χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία θα προέλθει από την Κομισιόν, η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αιτήσει των πολιτών, ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να προχωρήσουν για μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Ευχαριστώ. Μάλιστα και εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα η τελευταία ομιλία από τους εμπειρογνώμονες η Ντάγμαρ Ροτ Μπέρντ, πρώην Ευρωβουλευτής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πώς να συνδυάσω τώρα, πώς να περάσω από την ανάγκη να υπάρξει μια τέτοια κωδικοποίηση για ολόκληρη την Ένωση στις ανάγκες του δικού μας θεσμικού οργάνου, δικού μας λέω για την αποσυνήθεια του Κοινοβουλίου δηλαδή. Για να δούμε πού βρισκόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Αν συμφωνούμε ότι το διοικητικό δίκαιο είναι η βάση της δημοκρατίας για ασαφήνεια, για διαφάνεια και λόγω του δικαιώματος όσων επηρεάζουν οι νόμοι αυτοί να έχουν και αντιρρήσεις και προσφυγές, τότε αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κατάσταση. Πάντοτε βασιζόμαστε στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές επιλογές στην αντίδραση. Με κάποια ευχαρίστηση εξέτασα την κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 12 ο πρόεδρος του μου ζήτησε να εξετάσω πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, η συνδιοίκησή του. Μετά από μια έκθεση που είχα γράψει προηγουμένως για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, πράγματα όπως τη γαλάζιες κάρτες και την οφθαλμοθυρία, το Catch the Και όταν άρχισα να εξετάζω την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώς λειτουργούσε η διοίκησή του, ακόμη και για μένα μετά από τα 25 χρόνια εμπειρίας που είχα σε αυτό, που είχα ασχοληθεί με νομοθεσία για τα τρόφιμα και άλλα θέματα, Παρ' όλα αυτά με έκπληξη είδα πώς λειτουργούμε. Μερικά τα ήξερα, αλλά έμαθα και άλλα. Στα δυόμιση αυτά τελευταία χρόνια. Και είδα ότι αυτό που μας λείπει είναι η καλή διακυβέρνηση εδώ μέσα. Πρέπει βέβαια να μιλήσω προσεκτικά και ευγενικά, αλλά δεν υπάρχει καλή διακυβέρνηση. Πρέπει να το πω πολλές φορές το ανέφερα στο Προεδρείο προσπαθώντας να πω τα πράγματα θετικά, επικοδομητικά. Πρέπει όμως να το παραδεχτώ. Και επίσης παραδέχομαι ότι το η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι κλασική διοίκηση όπως στα Υπουργεία ας πούμε. Πρώτα λοιπόν είδα πώς λειτουργούν τα άλλα κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι υπάρχει πίσω τους, η λειτουργία τους, εθνικός κώδικας για τη διοίκηση. Παντού, στο Λουξεμβούργο, στην Αυστρία, παντού. Όπου υπάρχει εθνική διοίκηση, ε, ε, ε όπου υπάρχει εθνική διοίκηση, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνδυάσουμε την ιστορία και τις παραδόσεις 28-29 κρατών. Επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου πρέπει να συμπεριφέρονται σαν να έχουν διάφορα αφεντικά. Έχουμε εδώ ας πούμε τον κύριο Μπρέις, τον τμήματάρχη διοικητικό καθήκον, είναι διευθυντής, υπάρχουν οι γενικοί διευθυντές, ο γενικός γραμματέας. Εσύ όμως κύριε Σφόμποντα μπορείτε να θεωρείτε ότι εσείς είστε το αφεντικό του και όλοι από εσά, ο καθένας από εσά μπορεί να θεωρεί ότι είναι το αφεντικό του κυρίου Μπρέι. Αυτό το έλαβα υπόψη μου όταν εξέταζα αν λειτουργεί σωστά η διοίκηση του Κοινοβουλίου και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αρνητική απάντηση. Τα λέω γρήγορα γιατί ξέρω ότι θέλετε, ότι έχετε πίεση χρόνου λοιπόν. Σας υπενθυμίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα στον κανονισμό ως προς τα διοικητικά μόνο το άρθρο 222 που μιλάει για το Γενικό Γραμματέα και τη Γραμματεία και λέει ότι το Κοινοβούλιο θα υποβοηθιέται από το Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματεύς υπόσχεται στο Προεδρείο να, κάνει, να εκτελεί τα καθήκοντά του τελείως αδέκαστα. Είχε και κάνα δυο άλλα πράγματα, αλλά αυτό βασικά. Αυτό φυσικά δεν αρκεί. Και αυτό πιστεύουν και οι υπάλληλοι οι ευρωϊπάλληλοι. Μετά τις πρώτες άμεσες και καθολικές εκλογές του το 1979 υπήρχαν 1196 υπάλληλοι λιγότεροι από 2.000 και 5 γενικές διευθύνσεις. Ενώ στα τέλη του 2013 όταν τελείωσε η έκθεσή μου είχαμε 6.743 υπαλλήλους και 13 γενικές διευθύνσεις. Όταν εξελέγηνε εγώ το 89 για πρώτη φορά ήμασταν περίπου στη μέση. Άλλαξαν λοιπόν εκεί τα πράγματα πολύ. Η διαχείριση όμως, η, δι... η ικανότητα διαχείρισης αυξήθηκε, όχι δεν αυξήθηκε. Όταν μίλησα με ευρωυπαλλήλους εδώ και προσπάθησα να δω πώς λειτουργούν, ανακάλυψα κάτι που με εξέπληξε, ότι υπάρχουν δεκάδες κανόνων, εσωτερικών κανόνων από κάθε μονάδα, από τους διευθυντές, όπως ο κύριος Ιγκλέζιας εδώ, όπως ο Ρόμπερτ μπροστά μου, από γενικούς διευθυντές όπως τον κύριο Ντρέξλερ ή τον νομικό εμπειροχνόμονα Και όλοι αυτοί οι εσωτερικοί κανόνες μπορεί να καλύπτουν ή να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, αλλά είναι διαφορετικοί κανόνες. Σε κάθε γενική διεύθυνση ή διεύθυνση ισχύουν άλλοι κανόνες. Αυτό είναι περίεργο και ένας ευρωϋπάλληλος που είναι εδώ παρόν και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, η Διαμαρτίνες Ιγκλέσιας, προσπάθησε να ανακαλύψει πόσοι εσωτερικοί κανόνες εφαρμόζονται στο Κοινοβούλιο, τεράστια δουλειά γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες και έγραψε ένα τεράστιο έγγραφο που δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί αλλά θα δημοσιευτεί γιατί το ζήτησε το Προεδρείο από το Γενικό Γραμματέα δεν ξέρω αν είναι κανείς εδώ από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα σύντομα θα δημοσιευτεί ο κατάλογος που πρέπει να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του χρόνου λοιπόν τι είπα στο Προεδρείο ότι πρέπει να γίνει. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να είμαστε σαφείς για τις δομές. Στο Κοινοβούλιο λοιπόν το υψηλότερο όργανο είναι το Προεδρείο. Και θα έπρεπε αυτό να αποφασίζει τους γενικούς κανόνες τις γενικές αρχές, τις βέλτιστες πρακτικές στη διοικητική συμπεριφορά με επικουρικότητα τις ευθύνες, του συλλογικό χαρακτήρα και να τα λέει αυτά γραπτός και σαφώς. Οι βασικοί κανόνες της διοίκησης όπως η νομιμότητα, η αναλογικότητα, ο αδέκαστος χαρακτήρας, η ακαιρεότητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η εξυπηρέτηση των αναγκών του οργάνου. Αλλά είναι προφανής, αλλά χρειάζεται να εφευρεθούν και ορισμένα κανόνες που δεν υπάρχουν και που υπάρχουν σε άλλες διοικήσεις. Παραδείγματος χάρη το καθήκον να απαντάει κανείς ότι έλαβε κάποιο έγγραφο που του στείλανε. Αν μιλήσουμε και πάλι για το Γενικό Ρωματέα. Αν λάβει κάποιο σημείωμα από κάποιον, πρέπει το γραφείο του να απαντήσει «Ευχαριστώ, το έλαβα». Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη διοίκηση και απογοητεύσεις στη δουλειά της γραμματείας και των υπαλλήλων. Και έτσι χάνεται πολύ δυνατότητα και αξιοπιστία. Πρέπει επίση να υπάρχει το δικαίωμα να ακουστεί κανείς η ανάγκη να λαμβάνονται οι αποφάσεις με αναλογικό τρόπο και όχι και σύντομα και όχι να καθυστερούν οι υποθέσεις επί χρόνια. Ο κάθε υπάλληλο δηλαδή από κάθε μονάδα μέχρι το Γενικό Γραμματέα πρέπει να έχει γνώση όλων αυτών. Προσπάθησα να τα κάνω αυτά, να τα πω και όταν ήμουν βουλευτής, ελπίζω να κάποτε να εφαρμοστούν. Τώρα για τους γενικούς διαδικαστικούς κανόνες πρέπει να έχουμε άλλη προσέγγιση βασισμένη στην αποτελεσματικότητα. Παρακαλώ δώστε μου άλλα δύο λεπτά γιατί είχα πει ότι θα μιλούσα γερμανικά και τελικά αποφάσισα αγγλικά γι' αυτό τώρα ψάχνω τις εκφράσεις μου και καθυστερώ. Έπρεπε να είχα μιλήσει γερμανικά αλλά αφού οι περισσότεροι από εσάς δεν φορούσατε ακουστικά μιλούσατε ή καταλαβαίνατε αγγλικά το έκανα και εγώ. Συγγνώμη και για τις διερμηνήσεις. Τώρα, οι διοικητικές δομές λοιπόν. Οι κύριες ευθύνες για κάθε γενική διεύθυνση, για κάθε διεύθυνση, για κάθε μονάδα πρέπει να καθορίζονται από το Προεδρείο και να είναι γραπτά διατυπωμένες για το Γενικό Γραμματέα και τους Γενικούς Διευθυντές κτλ. Επίσης πιστεύω ότι το Προεδρείο πρέπει να αποφασίσει όπως στην Κομισιόν και σαφέστατα ότι ο Γενικός Γραμματέας και η... θα έχει συναντήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες με σαφές πρόγραμμα με τους υπόλοιπους γενικούς διευθυντές και διευθυντές από κάτω. Και διαφανώς. Αυτά προσπάθησα όλα να τα βάλω στην έκθεσή μου, αλλά φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβαν και ελπίζω, επειδή το Προεδρείο δέχτηκε την έκθεση, ότι κάποτε θα τα εφαρμόσει. Για την απλοποίηση των εσωτερικών κανόνων τώρα, όπως είπα, υπάρχουν αυτές οι δεκάδες εσωτερικών κανόνων και αναφέρονται σε ένα τρίστιλο έγγραφο που πρέπει να εφαρμοστεί υπομορφή εγχειριδίου καλής πρακτικής. Και ο πρόεδρος Σούλτς μου είχε ζητήσει να κάνω κάτι τέτοιο όταν ήταν δήμαρχος της μικρής του πόλης, βέβαια δεν του αρέσει να λέω ότι είναι μικρή αυτή η πόλη, αλλά είναι μικρή, έλεγε όταν ήμουν δήμαρχος είχα ένα εγχειρίδιο βελτίστων διοικητικών πρακτικών και ήλπιζα ότι θα υπάρχει και στο κοινοβούλιο, αλλά δεν υπήρχε. Τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και να δημοσιευτεί. Χρειάζεται επίση ενίσχυση των εσωτερικών κανόνων. Μερικοί είναι επικαλύψεις από άλλους και μπορεί να δοθεί διαφορετική λύση για το ίδιο πρόβλημα από διαφορετικές διευθύνσεις. Όσο για την νομιμότητα, όσοι είναι δικηγόροι όπως και εγώ, θέλουν όλα να δημοσιεύονται πριν εφαρμοστούν. Είναι και αυτό μια αρχή λοιπόν η δημοσίευση των κανόνων πριν εφαρμοστούν. Για μένα το Προεδρείο αυτό το έχει ήδη αποφασίσει, ε, γιατί δέχτηκε την έκθεσή μου. Είπαμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχουν όλα αυτά εφαρμοστεί και δημοσιευτεί. Δεν έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω να γίνουν πριν τελειώσει ο χρόνος για να μην χαραμιστεί και η δική μου δουλειά και του Λουίτζι Μπερλιγκουέρ. Όσοι ενδιαφέρεστε πάντως για τη διαφάνεια νομίζω ότι θα τα εκτιμήσετε όλα αυτά δεόντως ώστε να γίνει το όργανό μας πιο δημοκρατικό και να λειτουργεί καλύτερα και για τους πολίτες αλλά και για όλους εσάς και τους συνεργάτες σας. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου είναι πολύ καλή και της αξίζει περισσότερη δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας σχετικά με την δουλειά μας και τώρα ερωτήσεις. ενδεχομένως από τα μέλη προς τους διακεκριμένους ε, ομιλητές. Για χαόταλα. Μάλιστα ακούσαμε πολλά που μας εμπνέουν για αυτό το έργο το οποίο έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και καιρό. Υπενθυμίζω μια ιστορία όταν ο κ. Σιόντερμαν, ο πρώτος Ευρωπαίος Ομπουτσμαν ήρθε πριν από πολλά χρόνια εδώ στην Νομική Επιτροπή, χρειάστηκε να εξηγήσει τότε στην Νομική Επιτροπή ότι δεν θα ήταν και άσχημο οι Ευρωπαίοι δημόσιοι λειτουργοί να φέρονται σωστά στους Ευρωπαίους πολίτες. Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα περιοριστώ σε λίγες ερωτήσεις. Ακούσαμε από τον κύριο Χόφμαν ότι ίσως είναι ρεαλιστικό αυτό το διοικητικό δίκαιο να εφαρμόζεται στις διοικήσεις Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως σε αυτέ των χωρών μελών, ακόμα και αν εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Καταλαβαίνω αυτό το ρεαλιστικό, αλλά δεν θα οδηγήσει σε προβλήματα αυτό και σε νομικέ περιπλοκές και ποιε μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Δεύτερο, άκουσα ότι βασικό στόχος του εγχειρήματο θα πρέπει να είναι μια ενό είδου ολοκλήρωση και ενοποίηση των κατεσπαρμένων κανόνων και κωδίκων δεοντολογίας. Πώς όμως θα εντοπιστούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές στις οποίες θα βασιστεί το μελλοντικό αυτό Και μια παρατήρηση. Με ενθαρρύνει η προσέγγιση της αρμόδιας επιτρόπου κυρίας Γεωργίευα, γιατί μας είπε και στην ε, ακρόασή της ότι συνομιλεί με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τίμερμανς για το πώς θα αρχίσουν. Έχουμε λοιπόν πολλές ελπίδες για τούτη εδώ τη φορά ότι θα προκύψει κάποια πραγματική ουσιώδης πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι απευθυνθήκατε στον κύριο Χόφμαρ, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Βέβαια, οι χώρες μέλη όταν εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να ακολουθούν και μάλιστα είναι υποχρεωμένε να ακολουθούν τι βασικέ αρχέ του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα λέει αυτά η νομολογία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα έχει πει αυτά ξανά και ξανά στι αποφάσει του. Το άρθρο 41 πάντως τη συνθήκη είναι πολύ πιο περιοριστικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στην παράδοξη κατάσταση ότι οι χώρε μένουν υποχρεωμένε να εφαρμόζουν τι γενικέ αρχέ, αλλά με το 41 μπορούν να τα αφήσουν απ' έξω. Γι' αυτό θα είναι λογικό οι διοικητικές διαδικασίες να εφαρμόζονται και από τις χώρες μέλη όταν αυτές εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι λοιπόν θέμα προσέγγισης τόσο πολύ στη θεωρία, όσο του πώς θα διεξάγεται. Θα είναι πιο λογικό να αρχίσουν την ορθή πρακτική οι θεσμοί και ενδεχομένω μέσω της νομολογίας ή και μέσω της νομοθεσίας να προωθήσουν την, την ε, υιοθέτηση των αρχών αυτών ή να πούμε ότι ναι, από την αρχή αμέσω θα πρέπει να αρχίσουν οι ε, χώρες μέλη να εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο μαζί. Γι' αυτό είπα εγώ ότι υπάρχουν τόσοι τομεί όπου είναι κοινέ οι διαδικασίε και εκεί είναι αδύνατο να αφαιθεί η διακριτική ευχαίρεια στις χώρες μέλη εφαρμόζουν το εθνικό δίκαιο, διότι το αποτέλεσμα θα είναι μία ενιαία ε, διοικητική διαδικασία να βλέπει ότι μπορούν να εφαρμοστούν πολλές διαφορετικές αρχές. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο για τους πολίτες. Και βεβαίως είναι και αδύνατο για τα δικαστήρια να κάνουν μετά τη σωστή εξέταση των υποθέσεων. Γι' αυτό και πρέπει να ρυθμιστεί αυτό νομοθετικά. Ε, στι τομεί εκείνου όπου υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και ενό. Το δεύτερο που ρωτήσατε είναι σχετικά με τη μεθοδολογία. Πώ δηλαδή να εξευρεθούν οι βέλτιστε πρακτικέ. Αυτά τα πέντε χρόνια η ομάδα εργασία μα συνεργάστηκε με πολλού ειδικού από πολλέ χώρε μέλη, αλλά και άλλου εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάσαμε όχι μόνο τομεί πολιτική και τι έχει αποδώσει ω τώρα και μέσα σε ποια πλαίσια, αλλά και ποιε είναι οι παραδόσει των χωρών μελών. Αυτό μου φαίνεται λογικό ως προσέγγιση. Και εξ και όπως είπε και ο Λουίτζι Μπερλιγκουέρ, η ιδέα να εξετάσουμε πρώτα τα παραθυράκια, αυτό προτείνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε μα πού βρίσκονται κάποια κενά και να προσπαθήσουμε να βουλώσουμε τα κενά αυτά δεν είναι τόσο καλή προσέγγιση, διότι δεν μας επιτρέπει να δούμε την συνολική εικόνα και ιδίως τα μεγάλα ε, δομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη ποικιλομορφία των τομέων πολιτικής που οδηγούν σε αυτή την αδιαφάνεια του νομικού συστήματος. Και όταν μιλούμε για αύξηση της διαφάνειας και απλούστευση της νομοθεσίας, η πρώτη προσέγγιση θα πρέπει να είναι αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστερ έχει ένα ερώτημα. Θα ήθελα να σταθώ στη συζήτηση αυτή σε σχέση με το διοικητικό δίκαιο σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία για να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια το διοικητικό δίκαιο. Και δεύτερον, έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών για την Τσίτα και την TTIP. Η Κομισιόν όμως απέρριψε την ε, πρωτοβουλία αυτή λέγοντας ότι είναι μια διαδικασία εν εξέλιξη και επομένως η Κομισιόν δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει συνέχεια. Πρώτον λοιπόν, μήπως θα χρειαστεί μια διευκρίνηση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου για τις πρωτοβουλίες πολιτών και δεύτερον αν χρειάζεται μια διευκρίνηση των, ε, της σχέσης της Κομισιόν με τους ε, Ευρωπαίους ε, βουλευτές, γιατί οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές διεκδικούν την πρόσβαση στα έγγραφα διαπραγματεύσεων της TTIP και θα ήθελα να ξέρω η Κομισιόν με ποια ε, επιχειρηματολογία νομικού χαρακτήρα υποστηρίζει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτά τα έγγραφα και έχω καταθέσει και μια προφορική ερώτηση προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να έχω κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν για αυτό το σημείο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ε, πρέπει να αρχίσω εγώ, λέει η κυρία Ροτ Μπέρνετ. Ε, αυτό δεν έχει μεγάλη σχέση, πιστεύω, με το διοικητικό δίκαιο. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν διαθεσμικές συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων που έχουν συναυθεί και εγώ έπαιξα ρόλο στην ε, σύναψη μιας από αυτές τις συμφωνίες και στην περίπτωση αυτή η προσπάθειά μας ήταν να βρούμε μια ισορροπία, μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έγγραφα τα οποία έχουν διαβαθμιστεί ως εμπιστευτικά να μπορούν να τύχουν πρόσβασης. Αυτό είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Η διαφορά μας με την Κομισιόν στο παρελθόν πάντα ήταν το πώς διαβαθμίζεται ένα έγγραφο ως εμπιστευτικό ή ως απόρριτο. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε κανόνες ή είναι μια αυθαίρετη απόφαση της Κομισιόν. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με διοικητικό δίκαιο, είναι περισσότερο κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη διαθεσμική ισορροπία και τη σχέση των θεσμικών οργάνων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου με το Προεδρείο και τη Συνέλευση των Προέδρων και σε επαφή με τον πρόεδρο της Κομισιόν και τους άλλους επιτρόπους. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να διαπραγματευτεί μεταξύ αυτών των δύο φορέων. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν δεν έχει κάποιο ρόλο το διοικητικό δίκαιο. Το δεύτερο ερώτημα που θέσατε τώρα κύριε Κιώστερ είναι το κατά πόσον είναι σύνομο ή καλύπτεται από το διοικητικό δίκαιο η απόφαση της Κομισιόν η οποία μπορεί να απορρίψει μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία αναφέρεται σε μια ενεξελίξη διαδικασία. Εγώ τώρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό έχει να κάνει με το διοικητικό δίκαιο. Πρέπει να δούμε προηγουμένως ποιοι είναι οι κανόνες οι οποίοι διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ποιοι είναι οι κανόνες λοιπόν, πότε πρέπει να εγκριθεί και να δοθεί συνέχεια σε μια πρωτοβουλία πολιτών και πάλι αυτό καλύπτεται από μια διαθεσμική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και η Κομισιόν έχει δεσμευτεί για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να δώσει συνέχεια σε μια ε, τέτοια πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό θέλουμε εμείς με το διοικητικό δίκαιο και την ενότητά του να εξασφαλίσουμε τις περιπτώσεις αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν πολλές φορές με τρίτους, όπως είναι μια διαδικασία προσφορών, ένα πιλωτικό σχέδιο κτλ, που μπορούν να έχουν συνέπειες άχθους για τρίτους. Ε, στις περιπτώσεις αυτές όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα το διοικητικό δίκαιο που αναφέρθηκε. Πρέπει να βρούμε άλλες μεθόδου. Και εγώ θα μιλήσω λιγάκι στα γερμανικά. Το θέμα των πρωτοβουλειών πολιτών προφανώς είναι ένα θέμα του πώς πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία. Προφανώς μπορεί να υπάρξει μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία να ζητήσει μια δράση της εκτελεστικής εξουσίας. Οι περιπτώσει που αναφέρατε, η περίπτωση του TTIP είναι κάτι το οποίο πράγματι ενδιαφέρει την κοινωνία των πολιτών. Το θέμα τώρα των απορρίπτων πολιτών, ε, εγγράφων ή των εμπιστευτικών. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Το να ξέρει κανείς αν μπορούν τα έγγραφα αυτά να έχουν ένα τέτοιο χαρακτηρισμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πρόσβαση στην πληροφορία, όπως πάντα, είναι ένα κεφαλαιόδες στοιχείο της δημοκρατίας, της ε, διαφάνειας και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουν καταρχήν οι πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να γνωρίζουν τα εθνικά συστήματα, δεν ξέρουν το ευρωπαϊκό σύστημα και γι' αυτό είναι πιο σημαντικό να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Επομένω τα θέματα του διοικητικού δικαίου έχουν επίπτωση και στις σχέσεις με, τον πολιτο, με τους πολίτες. Το αν τώρα αυτά τα θέματα έχουν συγκεκριμένη συνάφεια ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία για την πρωτοβουλία των πολιτών. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί εδώ έχουμε ένα τομέα όπου υπάρχει μεν μια μερική ρύθμιση, η οποία βασίζεται εν μέρη στην ε, διαθεσμική συμφωνία, εν μέρη στη συνθήκη κτλ, αλλά η οποία αφήνει κάποια κενά και εκεί η ύπαρξη γενικών αρχών θα μπορούσε να επιτρέψει να καλύψουμε τα κενά αυτά. Γιατί φυσικά εδώ έχουμε να κάνουμε με την αρχή, με την απαρχή μιας διαδικασίας. Αλλά επίσης αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δείτε μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν την πρωτοβουλία αυτή. Δεν, δεν ξέρω τώρα αν το διοικητικό δίκαιο θα έπρεπε να μπαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως η πρωτοβουλία πολιτών, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν γενικές αρχές στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Τώρα δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει ήδη σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους τέσσερις διακεκριμένους ομιλητές μας. Ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχετε ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ για την έλευσή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να έχουμε και συνεργασία για τα θέματα αυτά και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. We continue with point number Πάμε στο σημείο υπαριθμών 5 που αφορά το εφικτό και το επιθυμητό του να μπορέσει η Κίνα να εμπνευστεί από το αστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Αν μπορώ να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις, προτού δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές μας και να παρουσιάσω την κατάσταση των πραγμάτων. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2014 η Ολομέλη έκλεισε την πρώτη ανάγνωση της πρότασης της Κομισιόν για τον λεγόμενο κοινό ευρωπαϊκό νόμο πολίσεων που είχε προταθεί από την Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2011. Πρόκειται για μια πρόταση κανονισμού που περιλαμβάνει κανόνες για το δίκαιο, για τις συμβάσεις πωλήσεων και που είναι μια ρύθμιση η οποία θα πρέπει να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα εθελοντικού χαρακτήρα εργαλείο το οποίο δεν αντικαθιστά το δίκαιο συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα συνεπάρχει ως ένα δεύτερο καθεστώς παράλληλα με το εθνικό δίκαιο και θα ισχύει μονάχα αν επιλέξουν οι συμβαλόμενες πλευρές να το χρησιμοποιήσουν. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει συντάξει μια εκτενή έκθεση αφού άκουσε τις απόψεις ε, των εμπλεκομένων σε ακροάσεις, σε ατελιέ, μαζί με ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους και εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων. Να καταγράψω επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η μονάδα για την εκτίμηση αντικτύπου έδωσε μια θετική γνωμοδότηση σε σχέση με την πρόταση αυτή. Η έκθεση ενεκρίθη στη Νομική Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013 και υπεστήριζε τον ε, προαιρετικό χαρακτήρα αυτού του εργαλείου και τη νομική μορφή ενός κανονισμού. Προτείνει ο κοινός, η κοινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πολίσεων να είναι διαθέσιμη σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια εξ δηλαδή μόνο τα ηλεκτρονικά συμβόλαια ουσιαστικά. Και η έκθεση αυτή διατηρεί την αρχή της ε, ελεύθερης επιλογής νομικών θεραπείων για τον καταναλωτή, αλλά απαιτεί μέσα σε δύο μήνες ο καταναλωτής να κοινοποιήσει την, ε, ε, την καταγγελία της ε, συνθήκης, της σύμβασης, από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο με το αγαθό το οποίο έχει αγοράσει. Και αυτά πέρασαν στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου του 2014 και η Επιτροπή μας έχει τώρα διορίσει τον Άλεξ Φως και την Αλεξάνδρα Μορέτη ως συνεισηγητές για τη δεύτερη ανάγνωση αυτού του νομοθετήματος. Αυτή η πρωτοβουλία η οποία είναι το επιστέγασμα ετών εργασίας και για την οποία η δική μας Επιτροπή έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο, πιστεύουμε ότι οι κινέζικες νομοθετικές αρχές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτό το νομοθέτημα και μετά από την επίσκεψή μας στην Κίνα ε, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τον κύριο Μέιερς, ο οποίος είναι συμβολιογράφος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία και επίσης καθηγητής στην νομική ε, σχολή του Πανεπιστημίου Σίγκουα στο Πεκίνο. Τον έχει προσκαλέσει να λάβει το λόγο ενώπιον της Επιτροπής μας σε σχέση με, την, με το εφικτό και την, το σκοπιμό του να δώσουμε τη δυνατότητα στην Κίνα να επωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Δίκαιο Πολίσεων. Θα, θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μέγε και μετά στον κύριο Σαντμάιρ από την Κομισιόν για να κάνει περαιτέρω σχόλια και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήματα. Δόκτωρ Μέγε, έχετε το λόγο. you, Chairman, Ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκλησή σα και για την εξαιρετική σας εισαγωγή του θέματο του σημερινού θέματος. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το πώς βλέπω τις δυνατότητες της διπυρωτικής συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και Κίνας. Όπως ξέρουμε και όπως είπα και στο έγγραφό μου, Αν δεν υπάρχει κάποια έλλειψη, κάποιο χάσμα μεταξύ νομικών συστημάτων, τότε μπορεί να, αυξηθούν οι εμπορικές συναλλαγές κατά 40%, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα θεμέλια, από τα θεμελιώδη κίνητρα της Ένωσης, αν αυξηθεί η εμπορική ροή κατά 40%. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ άλλων υπήρων. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αλλάζει τη θέση της. Όπως ξέρουμε και η υπηρετική Ευρώπη και η Κίνα έχουν σύστημα που βασίζεται στο αστικό δίκαιο αλλά τα τελευταία χρόνια Ο Αμερικανικός νόμος και οι νόμοι του Χονγκ Κόνγκ έχουν επηρεάσει πολύ την κινέζικη νομοθεσία. Και άρα το τωρινό νομικό σύστημα του αστικού δικαίου στην Κίνα είναι κάπως συγκεχημένο. Τι συνέβη. Έχουν πάρει κάπως ασύνδετα στοιχεία από το Αμερικανικό νομικό σύστημα, από το Ευρωπαϊκό νομικό σύστημα και τελικά το αποτέλεσμα είναι πολύ ασαφές και μεικτό. Πριν από μερικές εβδομάδες, τρεις εβδομάδες ακριβώς, έγινε το τέταρτο λέει ο μιλητής συνέδριο του Κομμουνιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Για πρώτη φορά το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, οι ηγέτες της Κίνας δηλαδή, δήλωσαν ότι ο νόμος είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων του συνεδρίου αυτού. Είναι από τα ανώτατα βήματα που μπορούν να συζητηθούν τέτοια πράγματα. Παράλληλα, οργανώθηκαν πολλές διεθνείς συναντήσεις στο πανεπιστήμιό μου στην Κίνα, Τσινκουά λέγεται, είναι πολύ δύσκολη η προφορά του, Τσινκουά, ε, όπου ήρθε και ένας από το Facebook, ο Ζικέρμπεργκ και μίλησε στους φοιτητές κινέζικα. Αλλά έγιναν και πιο βαρετές συνεδριάσεις με καθαρά νομικό περιεχόμενο. Και σε μία από αυτές ο αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου της Κίνας, ο δεύτερος αντιπρόεδρος, μας είπε ότι θεωρεί την τωρινή κατάσταση ως μία νομική άντιξη. Δημιουργούνται λέει νέα λουλούδια και μπορούν να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν της νομικής άνοιξης εγώ βλέπω σε διεθνείς διασκέψεις κλπ ότι η τωρινή νομοθεσία χωρίς να υπερβάλλουμε επικρίνεται από Κινέζους διανοούμενους και καθηγητές ιδιαίτερα σε αυτό το, για αυτό το αστικό δίκαιο το οποίο δημιουργείται τα τελευταία χρόνια. Χωρίς όμως επαρκές περιεχόμενο και σύνδεση μεταξύ των διαφόρων θεμάτων. Τι γίνεται λοιπόν. Μερικοί νόμοι επανεξετάζονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα, ξανααποτιμούνται, ο ε, εμπορικοί νόμοι, το αστικό δίκαιο και ...η δυνατότητα για την Ένωση να εξετάσει αν προγράμματα που έχει εκείνη εφαρμόσει από χρόνια δεν θα μπορούσαν να προταθούν και στην Κίνα, συζητιέται. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες βέβαια, δηλαδή η ιδέα της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης νομικών προγραμμάτων που έχουν εξεταστεί επαρκώς και έχουν αποδείξει την υψηλή τους ποιότητα σε ενωσιακό περιβάλλον, μήπως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλες αναδυόμενες χώρες και στην Κίνα. Αλλά είναι τέτοια η συγκυρία ώστε αυτή η νομική άνοιξη που αφορά μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, εάν βασιστεί συμβατή, αν γίνει συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό νέες τεράστιες δυνατότητες και για τις δύο οικονομίες και για την ευρωπαϊκή. Θα έλεγα ότι η ιδέα αυτή δεν αφορά μόνο επιτυχίες όπως το σχέδιο CESL, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υπάρξει και προγράμματα, σχέδια από την Ευρώπη που θα έλεγα ότι απέτυχαν τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου. Αυτό μπορεί να συνέβη για πολιτικούς λόγους, μπορεί μερικά προγράμματα να ήταν υπερβολικά φιλόδοξα, αλλά παρόλα αυτά τα σχέδια και προγράμματα που απέτυχαν μπορούν και αυτά να είναι πηγή έμπνευση για άλλες χώρες. Και η ιδέα αυτή ότι μπορεί κανείς να συνδυάσει τη βάση νομικών συστημάτων μεταξύ τους είναι κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα ή σχέδιο που το ενέπνευσε την ιδέα έχει πετύχει ή αποτύχει. Διότι πάλι θα βοηθούσε στην συμβατότητα των νομικών συστημάτων. Τέλος θα έλεγα ότι οι Κινέζοι ακαδημαϊκοί που συνάντησαν... είναι ενθουσιώδεις για το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα και θεωρούν ότι είναι πολύ σοφή η ιδέα της επικουρικότητας Όταν μιλάω για, και παρουσιάζω, κάνω παρουσιάσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Κίνα, μου λένε καμιά φορά ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να μας δώσουν κατευθύνσεις όχι σαν διαταγές αυτοκρατορικές αλλά κατευθύνσεις Και για να καταλήξω τελικά πάλι, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την Ευρώπη ώστε να αποτελέσει έμπνευση και για άλλα νομικά συστήματα και χώρες και για πολλούς λόγους η Κίνα θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σταντμάιερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ. Για να μιλήσω για τη δυνατή μεταλαμπάδευση του ευρωπαϊκού δικαίου πολίσεων στην Κίνα. Η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα. Υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες του Ειρηνικού και της Ασίας που από ό,τι γνωρίζουμε ενδιαφέρονται να αναθεωρήσουν ή να μεταρρυθμίσουν τον νόμο περί συμβάσεών τους. Η Ιαπωνία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και φυσικά και η Κίνα. Η άποψή τους είναι ότι θέλουν να προσαρμόσουν το, την νομοθεσία πολίσεών τους καλύτερα προσαρμοσμένη στα θέματα παγκοσμίου εμπορίου. Γι' αυτό κοιτάζουν πρώτα προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ή για ήπια νομοθεσία όπως είναι διεθνείς ε, ε, συμφωνίες και για το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Αλλά κοιτάζουν επίσης και στο, στην νομοθεσία των κύριων εμπορικών εταίρων τους για βέλτιστες πρακτικές και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωπαϊκοί νόμοι και αυτό έλαβαν και την εθνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την δυνατότητα να τύχουν εξαγωγής προς την ε, Κίνα ή την περιοχή του Ειρηνικού. Ο κοινός, η κοινή νόμη περί, η κοινή μάλλον νομοθεσία περί πολίσεων μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Γιατί υπάρχει καταρχήν ένα εκτατικό, ένα εκτενές πλαίσιο συγκριτικού δικαίου, το οποίο βασίζεται στις πρακτικές όλων των κρατών μελών, αλλά και το οποίο βασίζεται και στο κοινοτικό κεκτημένο και βασίζεται βέβαια και σε διεθνή νομικά εργαλεία όπως είναι η Σύμβαση της Βιέννης για την πώληση αγαθών και την, ε, τις αρχές της Ινιτρουά. Και η βασική αρχή λοιπόν είναι να υπάρξει ο συνδυασμός των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων αφενός και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών αφετέρου. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά επιτελείται και μια μεταρρύθμιση του δικαίου καταναλωτών. Είναι λοιπόν μια πηγή εμπνεύσεως το, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Μάιερ και αυτό το οποίο είπε μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πρόκειται για αυτοκρατορικό διάταγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο Ευρωπαϊκός Νόμος Περιπολίσεων έχει στο επίκεντρό του την επιλογή. Δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παρέμβουν στην ε, μακροχρόνια παράδοσή τους σε σχέση με, τον, το δίκαιο των συμβάσεων, αλλά είναι μια πρόσθετη επιλογή η οποία παρέχεται τόσο στους πολιτές όσο και στους ψωνιστές και τους καταναλωτές συγκεκριμένα για να μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις διαμεθοριακές τους συναλλαγές. Κάτι το οποίο θα πράξουν μόνο αν για αυτούς υπάρχει κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο μπορούν να προσποριστούν. Για τον πολιτή λοιπόν σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μειώσει το κόστος συναλλαγών γιατί μπορεί να πολύ επί τη βάση ενός μονάχα δικαίου και μιας πλατφόρμας πληροφορικής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγοραστή σημαίνει ότι θα έχει ένα ευρύτερο φάσμα προμηθευτών, περισσότερα προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές ε, τιμές και σε επίπεδο καταναλωτή θα υπάρχει μια ε, εναρμονισμένη προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και θα υπάρχει παντού κάτι το οποίο θα είναι παρόμοιο με το εναρμονισμένο πλαίσιο ή, βελτι, βέλτιον. Επομένως δεν πρόκειται για μια αυτοκρατορική διαταγή. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο συμφέρον να προωθήσει αυτή την νομοθεσία για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς. ότι τέτοιοι λόγοι είναι ότι αν εμείς ως ε, σημαντικός εμπορικός εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σύγκληση στα θέματα αυτά, αυτό σημαίνει για τις δικές μας επιχειρήσεις υποδέστερο κόστος. Εάν επίσης μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για τους εμπορικούς εταίρους μας να υιοθετήσουν κάποια τμήματα της δικής μας νομοθεσίας, αυτό είναι πραγματικά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις δικές μας επιχειρήσεις έναντι αυτών των Αμερικανών, πουχού. Είναι σαφές όμως ότι και για τους νομομαθείς οι οποίοι δίδουν νομικές συμβουλές στους πελάτες τους για τι εξαγωγέ και σε αυτού οι οποίοι συμμετέχουν σε διεθνή διατητικά δικαστήρια, το να υπάρχει αυτή η ενότηση. Επομένω, για όλου αυτού του λόγου, εμεί μπορούμε να κερδίσουμε μονάχα από το να κάνουμε τι προσπάθειε εξαγωγή τη νομοθεσία μα. Αυτά ήθελα να σα πω λοιπόν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε την έγκριση αυτού του κοινού ευρωπαϊκού νομοθετήματος για τις πωλήσει και να ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να ανθίσουν χίλια κινέζικα νομικά λουλούδια με τον νόμο αυτό. Uh, uh, είπα πριν ότι είστε από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλλον δεν το είπα και το λέω τώρα. Τώρα λοιπόν έχει έρθει η ώρα να θέσετε ερωτήσεις, mm. κύριε Ευρωβουλευτέ και κυρίες Ευρωβουλευτέ. Κύριε Μουρίνιο Πίντου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Με μεγάλη χαρά καταγράφω το ενδιαφέρον της Κίνας για την Ευρωπαϊκή Εμπορική Νομοθεσία που είναι εξάλλου μια πολύ εξελιγμένη σε τεχνικό επίπεδο νομοθεσίας. Θυμάμαι τις πρώτες προσπάθειες για την κωδικοποίηση της εμπορικής νομοθεσίας τον κώδικα του Ναπολέοντος στις αρχές του 19ου αιώνα. Θα ήθελα όμως να γνωρίσω και γι' αυτό θέλω να θέσω το ερώτημα. Είναι το ενδιαφέρον της Κίνας μόνο για την εμπορική νομοθεσία ή ενδιαφέρεται για άλλους τομείς νομοθεσίας όπως πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, η εγγυήσει των δημοσίων ελευθεριών, η προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών έναντι της κρατικής εξουσίας και η αρχή, οι αρχές της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κτλ. Δεν ε, ξέρω και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την Κίνα και σε αυτά τα επίπεδα και άλλες περιοχές του κόσμου ή αν τελικά όλα αυτά συμποσούνται μονάχα στα θέματα κίνησης των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων και του χρήματος και τίποτα παραπάνω. Θα συγκεντρώσουμε μερικά ερωτήματα πρώτα και μετά θα ζητήσουμε να απαντήσετε. Ποιος? Μας λέτε σήμερα ότι η Κίνα θαυμάζει το εμπορικό μας δίκαιο ή ότι το θεωρεί θετικό και για εκείνη, την επικουρικότητα, ότι δεν πρόκειται για αυτοκρατορικά διατάγματα, όλα αυτά είναι λίγο εκπληκτικά ως αποτίμηση εκ μέρους της Κίνας που δεν έχει τη φήμη πολύ εύκαμπ του κράτους. Μπορούμε να χαρούμε και εμείς για τις οικονομικές προοπτικές που μπορεί να φέρει αυτή η έμπνευσή μας προς την Κίνα αλλά δεν ξέρουμε αν η Κίνα δεν θα δώσει τελικά προτίμηση στο αμερικανικό σύστημα. Υπάρχει όμως και κάτι αρνητικό. Δεν είναι εκπληκτικό ότι η Κίνα μας εγκρίνει σε εισαγωγικά, ενώ η ίδια δεν είναι κανένα υποδειγματικό κράτος όλα τα συγχαρητήρια που μας δίνει η Κίνα μου φαίνονται λίγο ανησυχητικά. Τι νομίζετε κι εσείς. Χάουταλα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Μάγερ για τη νομική άνοιξη της Κίνας. Ίσως πρέπει να δούμε τη συνεργασία σε τομείς, σε διάφορους τομείς στην Κίνα γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δούμε σε ποιες αρχές βασίζεται. Πέρα και από το θέμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ξέρουμε ότι υπάρχει νομική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών και Κίνας από χρόνια και ότι Προσπαθήσαμε να εξαγάγουμε τις ιδέες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν υπήρξε και πολύ επιτυχής η προσπάθεια αυτή. Ίσως υπάρχει και άλλος τρόπος να τα δούμε όλα αυτά. Ας πούμε να διασφαλιστεί ότι ο πολίτης θα έχει κάποια θέση, αν και πρόκειται για συλλογικού χαρακτήρα κυρίως διαδικασίες στην Κίνα. Ίσως όμως ο πολίτης να μπει κάποτε στο κέντρο, γιατί μου φαίνεται ότι Προς τα εκεί τα πράγματα και θα έπρεπε να το δούμε. Dr. Myers, you have the Ο Δόκτωρ Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μ' άρεσαν πολύ οι ερωτήσεις. Διότι εγώ βασίστηκα και θεωρητικά και πρακτικά στα νομικά πρόσωπα και πάντα λέω στην Κίνα ότι τα νομικά πρόσωπα και το επιχειρηματικό δίκαιο εν μέρη είναι μια μεταφορά. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για νομικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνάψουν συμβάσεις, να αποφασίσουν ελεύθερα, τότε έχουν κάποια θέση. Και αυτό το μήνυμα ακούγεται, περνάει. Ιδιαίτερα για το τρίτο ερώτημα θα ήθελα να πω ότι κατάλαβα ότι μπορεί να υπάρξει και έμεση προσέγγιση, δεν είναι ανάγκη να γίνει άμεση κατά μέτωπον αντιμετώπιση. Ο έμεσος τρόπος μερικές φορές είναι πιο βιώσιμος και πιο επιτυχής από ότι αν επιμείνει κανείς κατά πρόσωπο με ορισμένες αξίες που θέλουμε να τονίσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να αρχίσουμε από πρακτικά πράγματα όπως τα κεφάλαια και οι επιχειρήσεις και ελπίζω ότι με έξυπνο τρόπο, αν κρατήσουμε τη στρατηγική μας καθαρή, θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσω των κεφαλαίων και των επιχειρήσεων και να περάσουμε και άλλες αξίες. Κανένα σχόλιο. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ ο καταλληλότερος να μιλήσω για θέματα εξωτερικής πολιτικής με την Κίνα. Αλλά εδώ μιλάμε με βάση αυτά βασικά που είπε η κυρία Χάουταλα, δηλαδή με βάση το συμβασιακό δίκαιο που είναι η βάση του ευρωπαϊκού δικαίου για τις πωλήσει και τα εμπορικά. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική βάση. Δεύτερον, οι ευρωπαϊκοί αυτοί νόμοι βασίζονται σε συμφωνίες, δεν επιβάλλονται σε κανέναν, μόνο αν οι συμβαλόμενοι δέχονται, θεωρούν ότι υπάρχει πλεονέκτημα. Και το τρίτον, σίγουρα πολύ μεγάλο ψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή υπονοείται επίσης, δηλαδή προστασία του πιο αδύνατου μέρους Αφού μιλάμε για αξίες και αν πρέπει έμεσα όπως είπε ο Δόκτωρ Μάγερ να περάσουμε τις αξίες αυτές στην Κίνα μπορεί έτσι να βγει κάτι θετικό. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την παρατηρήσή σας. Παρατήρησή σας. βέβαια σπούδασα τα νομικά μου προ 35 ετίας υπό απολυταρχικό καθεστώς και ο πρώτος ορισμός δικαίου που άκουσα είναι ότι ήταν εργαλείο του αγώνα της ε, εργατικής τάξης. Τελεία. Αυτό είναι όλο. Έτσι λοιπόν εκτιμώ ιδιαίτερα το ενδεχόμενο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων να έχει κάποια θετική επιρροή στο Κινέζικο Δίκαιο. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις, ούτε κανένα να γύρει την χείρα Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ενημέρωση και θα διακόψω τώρα την συνεδριασή διότι το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν όλους όσοι δεν δικαιούνται να παρίστανται να αποχωρήσουν.